Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα προβλέπεται η πολύ ευχάριστη συνάντηση με τον γερουσιαστή Τζον Χόγκ, πρόεδρο της Γερουσίας της Αυστραλίας, ο οποίος θα μας κάνει μια εισήγηση ως προσχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Όπως γνωρίζουμε, το γεγονός μαζί, το ότι μαζί μας ε, βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος Ρόμπερτ Στέρντι της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου δείχνει τη σημασία των ε, σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Δεν μιλάμε μόνο όμως για εμπορικές σχέσεις που μας συνδέουν Μιλάμε για κοινέ αξίες και μία παρόμοια θεώρηση του κόσμου. Έχουμε διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν, αναφέρομαι σε μερικά μόνο. Την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέματα ασφάλειας και άμυνας, συνεργασία στους πολυμερείς οργανισμούς και το βασικό ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. Όλοι γνωρίζουμε το στρατηγικό ρόλο της Αυστραλίας στα πλαίσια της Ανατολικής Ασίας πράγμα που μας οδηγεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεώρηση για το τι ε, συμβαίνει σε εκείνη την πλευρά του κόσμου. Και Στη συνέχεια, πολλοί βουλευτές θα απευθύνουν το λόγο και ερωτήσεις στον γερουσιαστή, στον πρόεδρο της Γερουσίας. Θα δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο, τον κύριο Στέρντι, για έναν θερετισμό, χαιρετισμό, αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να καλωσορίσω και εγώ τον γερουσιαστή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα η επίσκεψή σας μέχρι τούδε. Ήμουν πρόεδρος ε, της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας και η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν έκτοτε μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας μπορούμε να επεμβαίνουμε στην τελική μορφή της συνθήκης και ολόκληρο το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της συναπόφασης. Χαίρομαι λοιπόν γιατί προσήλθατε σήμερα στη σημερινή μας συνάντηση και ορισμένα από τα θέματα που μας απασχολούμε στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου και θα ήθελα να ακούσω με ενδιαφέρον την άποψή σας σε σχέση με τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σε σχέση με το γύρο της Δόχα. Πολλοί είμαστε Απογοητευμένη. Εγώ πιστεύω στις πολυμερείς και όχι τις διμερείς συμφωνίες μέσα στα πλαίσια του αναπτυξιακού αυτού γύρου και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που το χρειάζονται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, λοιπόν, έχουμε μια πλήρη στρατηγική, μια πλήρη υποστήριξη. Και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε σαν σχέδιο Β τη στιγμή που ο γύρος της ε, Ντόχα πλέον έληξε, έληξε άδοξα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε διμερείς σχέσεις με την Αυστραλία, τώρα εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε και οι εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες της κοινοπολιτείας να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε τις διμερείς συμφωνίες, προβλήματα στις εμπορικές, στις εμπορικές συμφωνίες, τι βλέπετε σε σχέση με μέσα διαφύλαξης των εμπορικών συμφωνιών. Και θα παραμείνω εδώ επί του παρόντος. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και ας αφήσουμε το λόγο στον γερουσιαστή, τον πρόεδρο της Γερουσίας, στον κύριο Χόγκ. Θα σας ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον κύριε Χόγκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για το θερμό σας καλωσόρισμα και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω έρθει πρώτη φορά πέρσι με την ίδια ιδιότητα ο πρόεδρος της Γερουσίας και αυτή είναι η δεύτερη φορά. Ε, θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο και όχι την εκτελεστική πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό το λέω σαφέστατα εξ αρχής έτσι ώστε να καταλάβουν οι συνομιλητές μου ότι έργο μου είναι να εξασφαλίσω τις σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλίων και να τις ενισχύσω και ενθαρρύνω μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κοινοβουλίου της Αυστραλίας. Πολλοί ε, πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι εύκολο, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Σαφώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε υπουργικό επίπεδο και σε ηγετικό επίπεδο μεταξύ ηγετικών στελεχών. Δεδομένου ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση όμως το επίπεδο το κοινοβουλευτικό, στο επίπεδο των νομοθετών εκεί παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, ανταλλαγής απόψεων και έτσι να βοηθήσουμε τις κοινέ διαβουλεύσεις ως νομοθέτες. Πριν από 8 εβδομάδες καλωσόρισα μία αντιπροσωπεία στην Αυστραλία ε, με την ευκαιρία της 30ης επαιτίου των σχέσεων της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η σημασία αυτών των σχέσεων έχουν αναβαθμιστεί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και χάρηκα ιδιαίτερα που ακούστηκε αυτό ευθύ εξ αρχής. Αναγνωρίζουμε τώρα, όχι βέβαια ότι κάτι έλειπε από την ε, ημερήσια διάταξη μας ε, στις ε, σχέσεις μας, αλλά αναγνωρίζουμε πόσο ακόμα περισσότερο σημαντικές είναι οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στέλνουμε ένα μήνυμα σε εσά για μια αλλαγή προσέγγισης στην κυβέρνηση με τον τρέχοντα πρέσβη μας, τον κύριο Νέλσον και αυτή η αλλαγή της σχέσης ε, δείχνει ότι θέλουμε να ε, ε, εντείνουμε ακόμα περισσότερο, να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και στο μέλλον. Βεβαίως συμμεριζόμαστε πολλές κοινέ αξίες. Σωστά ελέγχθη αυτό. Περισσότερα στοιχεία μας ενώνουν από ότι μας χωρίζουν και στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας ε, αναπτύσσουμε συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος, αλλαγής κλίματος, εμπορίου αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί στενά μαζί μας σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Ασία. Σαφώς, θεωρούμε τον εαυτό μας τμήμα της Ασιατικής Υπήρου και θεωρούμε ότι είμαστε και ότι συμμετέχουμε ε, μακροπρόθεσμα στις ασιατικές εξελίξεις. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ σημαντική σχέση με την Κίνα επί μακρό χρονικό διάστημα τόσο ευρεία σχέση μάλιστα που πριν από δύο χρόνια και λόγω αυτής της στενής σχέσης που έχουμε με την Κίνα και έτυχε τότε ε, να είμαι πρέσβης ε, της ε, Αυστραλίας στην Κίνα δέχτηκα, μπόρεσα να οργανώσω μία επίσκεψη Αυστραλών βουλευτών στο Σιβέτ. Ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκε μία επίσκεψη Αυστραλών βουλευτών στο Σιβέτ. Αυτό το γεγονός δεν ήταν ασήμαντο, ήταν ε, σημαντικό διότι υπήρχαν ορισμένα ευαίσθητα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και ορισμένα έντονα προβλήματα πριν από μερικούς μήνες, πριν από την επίσκεψη. Αυτό δείχνει λοιπόν πόσο στενές είναι οι σχέσεις μας και με αυτή την περιοχή του κόσμου αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, δεν είναι η σχέση μόνο αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια, είναι μια συλλογική συνεργασία. Είναι μια συνεργασία που βασίζεται και σε διμερείς σχέσεις που έχουν εδρεωθεί εδώ και πολύ καιρό. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτές τις διμερείς σχέσεις όπως φάνηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες που επισκέφθηκα τη Σουηδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Και δεν προσπαθούμε να προωθήσουμε μόνο ε, σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης τις σχέσεις μας, αλλά να πτήσουμε ταυτόχρονα και τις διμερείς. Στο θέμα του εμπορίου, συνήθως ε, αυτό το θέμα είναι στην, ε, το αναπτύσσει ο υπουργό Εμπορίου, ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος και γνώστης των θεμάτων, αλλά μπορώ αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ να αναλάβω αυτό το ρόλο και εγώ ε, και να πω ότι και στο εμπορικό πλαίσιο πάντοτε Προσπαθούμε να ε, δείξουμε ότι ο γύρος της Ντόχα ήταν μια επιτυχία, ήταν επιτυχής. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι εάν θέλουμε το μέλλον μας ε, να είναι εξασφαλισμένο όχι μόνο στην στον οικονομικό χώρο στην Αυστραλία και γύρω από την Αυστραλία αλλά παγκοσμίω, τότε το θέμα του ελευθέρου εμπορίου πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα διότι αλλιώς η ανάπτυξη θα σταματήσει, θα κολλήσει και θα δημιουργήσουμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Πάντοτε ήμασταν πρωτοπόροι ε, στην προσπάθεια απελευθέρωσης του εμπορίου εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Η επιλογή την οποία εμείς προτιμούμε ήταν πάντοτε να στηριχθούμε σε πολυμερή ε, ε, σώματα, σε πολυμερείς οργανισμούς και συμφωνίες και όχι σε διμερείς. Και γιατί, διότι σε πολυμερείς οργανισμούς μπορούμε να ε, συνάψουμε ορισμένες εμπορικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου πολύ ε, καλύτερα από ό,τι σε διμερή βάση. Όποτε ξέρετε, αντιμετωπίζουμε τώρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και αυτό έχει επηρεάσει ε, και την Ευρώπη και μας. Έχουμε επενδύσει σε ένα πακέτο κινήτρων και αναζωγόνησης της οικονομίας. Όχι όμως υποφέρουμε και εμείς από ύφεση παρόλο το πακέτο αυτό. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον με αυ- εν ώψη της παγκόσμιας κρίσης μπορέσαμε να, να αποφύγουμε τον πάτο, δηλαδή το, τη χειρότερη πτυχή της οικονομικής ε, κρίσης. Αυτό το πακέτο λοιπόν δεν μας έσωσε τελείως αλλά μπόρεσε να μας βοηθήσει. Ε, να βγούμε, να βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση. Επίσης η συναλλαγματική μας ισοτιμία είναι ευμενής, έχει εξελιχθεί καλά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία ε, Αυστραλίας-Ευρώ διότι η γυναίκα μου έτσι ξοδεύει λιγότερα χρήματα από την τσέπη μου όταν ψωνίζει εδώ. Έχουμε λοιπόν ωφεληθεί σε αρκετά σημεία. Η παγκόσμια οικονομία έχει αρχίσει να βελτιώνεται δραματικά. Θέλουμε να αναπτυχθεί περισσότερο η απελευθέρωση του εμπορίου και των αγορών. Η απάντηση είναι ναι διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε την απασχόληση που χρειάζεται για να καλύψουμε την υποχρέωση που έχουμε στους πολίτες μας να ζουν με αξιοπρέπεια, με αυτοπεποίθηση και να συμμετέχουν στην οικονομία της Αυστραλίας. Αυτό το οποίο χρειάζεται ε, με τις παρούσες συνθήκες είναι να βοηθήσουμε τη μετάβαση από το καθεστώς στο οποίο βρισκόταν η βιομηχανία και το ε, καθεστώς, το οικονομικό κλίμα αν θέλετε, όπως ήταν στο παρελθόν, να μετακινηθούμε προς μια νέα εποχή όπου θα δρέψετε τους καρπούς των ε, διαπραγματεύσεων, των επιτυχών διαπραγματεύσεων. Ένα από τα θέματα τα οποία εμείς θέτουμε πάντοτε στο τραπέζι, σε οποιαδήποτε εμπορική διαβούλευση, είναι το θέμα των αγροτικών προϊόντων. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ιδίω σε σώματα, όσο σε οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε θεσμικά όργανα. Μία λοιπόν που έσυξε το θέμα αυτό και ξέρω ότι θα μου θέσετε ερωτήσεις, τις οποίες ελπίζω να, απαντήσει, να απαντήσω. Να πω ότι εμείς στο κοινοβούλιο μας έχουμε μία κοινή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που καλύπτει και τα δύο σώματα μέλη και από τη Γερουσία και από το Κοινοβούλιο και εξετάζει, μελετάει ε, πολλά θέματα μεταξύ των οποίων άμυνα, εμπόριο και ιδίω ανθρώπινα δικαιώματα. Nothing Και ε, επικεντρώνουν την, την προσοχή τους σε αυτή η μεικτή επιτροπή σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία συζητούμε με πολύ προσοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι σας ε, κατανοήσατε πόσο μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και με τι ενδιαφέρον αναμένουμε τις συζητήσεις μας με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, διεξοδική παρουσίαση, αν και συνοπτική. Τώρα ανοίγει η συζήτηση, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις. Ο πρόεδρος Χόγκ είναι στη διάθεσή μας για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις ή να ακούσει τη σκέψη σας. Ο κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Στα αγγλικά. Α, έπεσε ένα νερό. Εντάξει, δεν είναι και κανένα τεράστιο σεισμό. Σα ε, Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα ε, το οποίο δεν θίξατε στην εισαγωγή σας, αλλά ήταν στην ημερήσια διάταξη και με διέφερε εδώ και χρόνια συμμετέχω και στην Ισομερή Συνέλευση και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, εκεί παίζει ρόλο κλειδί ο ειρηνικός και χαιρόμαστε πάρα πολύ ε, που και εσείς κάνετε προσπάθειες σταθεροποίησης ε, στον ειρηνικό όπου υπάρχουν πάντα αιστείες ανάφλεξης στα νησιά Φίτζη, ε, γίνονται κατά καιρού πραξικοπήματα ή Σολομών νήσους. Ε, το 2005 νομίζω στείλατε μια ειδική αποστολή εκεί για να αντιμετωπιστεί η κρίση και άλλα μέρη στον Ειρηνικό όπου επικρατεί ένταση. Εσείς πώς ε, αξιολογείτε την εξέλιξη στα Φίτζη, στην ίσο του Σολομόντα, έχει επιπτώσεις ε, στη μετανάστευση για σας αυτό, στην περιφερειακή πολιτική εν Και επειδή έχουμε χρήματα ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη για τις χώρες αυτές, πού θα βλέπατε μεγάλες δυνατότητες ε, συνεργασίας για να πιάσουν τόπο τα χρήματά μας. Και ευχαριστώ. Ο κύριος παρακολουθήσαμε εκ του uh, to ο, η απάντηση του Προέδρου της Γερουσίας. Πάντα είχαμε πολύ καλές ε, σχέσεις με αυτές τις ε, χώρες προς βοράν και βόρειο-ανατολικά και βορειοδυτικά. Σε σχέση με τις νήσους Φίτζι, Δεν θέλαμε να επιβάλλουμε καμία λύση εμείς. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με τις χώρες του νοτιοδυτικού ειρηνικού για να δούμε κατά πόσο τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν ειρηνικά. Δεν θεωρούμε ότι εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε επικεφαλής ενός τέτοιου εγχειρήματος, για να το θέσω έτσι. Συνεργοζόμαστε εκ του σύνεγγης με την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, έτσι ώστε να έχουμε μία αγαστή σχέση. Έχουμε αυξήσει τη βοήθεια, την υπερπόντια βοήθεια, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες σε θέματα διακυβέρνησης και κράτους δικαίου καθώς και πρωτογενείς υπηρεσίες, χορήγηση πρωτογενών υπηρεσιών ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του AIDS. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα ως προς την Παπούα Νέα Γουινέα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και γνωρίζω ότι πολύ συχνά δεχόμαστε πολίτες από χώρες όπως τα νησιά του Σολομόντα, καθώς και άλλες χώρες που γνωρίζουν μεταβατικές κυβερνήσεις. Uh, than... Ιδιαίτερα στα πλαίσια της δημοκρατίας του, της Τόγκα που γνωρίζει μια μεταβατική κυβέρνηση και από όσο ε, γνωρίζω υπάρχουν εξελίξεις και Στις 25 Μαΐου θα μεταβώ στην Τόγκα έτσι ώστε να συζητήσουμε για την εφαρμογή μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν θα κάνω κανένα κήρυγμα, δεν θα τους πω τι πρέπει να κάνουν. Εκείνοι ήρθαν σε μας, παρατήρησαν πώς λειτουργούμε και εμείς θα μεταβούμε εκεί γιατί θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στους πολίτες. Είμαστε πολύ δραστήριοι σε όλη την περιοχή και στην Ινδονησία γιατί ε, εφόσον πρόκειται για μια μεγάλη χώρα, γείτονα χώρα, δεν μπορούμε παρά να έχουμε καλές σχέσεις. Και εδώ τίθεται και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, που γνωρίζω ότι αντιμετωπίζεται, ότι αποτελεί δυσκολία και για σας και, μας, και για μας ισχύει το ίδιο. Και θα ήθελα να πω ότι ως προς την Παππούα Νέα Γουινέα, και τις χώρες του νοτιοδυτικού ειρηνικού. Δεν προέρχεται από εκεί ε, αυτό το ρεύμα, αλλά από, το, από βορειοδυτικά, από τη Μαλαισία δηλαδή, την Ινδονησία και μετά έρχεται σε εμάς. Βεβαίως, δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις με τις μεταναστευτικές ροές στη Λαμπεντούζα ή στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα ύψιστο ζήτημα ανθρωπιστικής υφής και μας δημιουργεί δυσχέρειες. Δεν ξέρουμε πώς και εμείς να αντιμετωπίσουμε τους παράνομες μετανάστες που έρχονται στις ακτές μας. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας. abbiamo ora un intervento di un collega della Commissione Commercio Internazionale. Ο κύριο Σόλτς έχει το λόγο από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε δύο σημεία. Και αυτό... Εδώ είμαι. Που είπε ο κύριος Ρόμπερτ Σέρντι, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής μας στην αρχή. Και ε, σας ερωτώ πώς εκτιμάτε την προοπτική και τις εξελίξεις ε, τις πραγματικές του γύρου του Ντόχα. Είναι ρεαλιστικό στόχος για την Αυστραλία να εμπλακεί εκεί και πώς εμπλέκεται σήμερα ε, στις διαπραγματεύσεις που είναι αποφασιστικές για να οδηγηθεί σε κάποιο πέρας ο γύρος της Ντόχα. Και εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει προθυμία μεταξύ των εταίρων, ιδιαίτερα των επιτυχμένων βιομηχανικών κρατών, να κάνουν κάτι για να ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα. Η δεύτερη ερώτηση συνδέεται λίγο με την προηγούμενη. Συζητούμε για πολυμερή περιφερειακή ε, εμπορική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με περιφερειακούς οργανισμούς και είναι δεδηλωμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εστιάζεται εκεί και να μην μπαίνει στον πειρασμό να κάνει διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Γιατί έχουμε, θα το χαρακτήριζα μέχρι και πληθωρισμό σήμερα τέτοιων διμερών εμπορικών συμφωνιών. Εσείς που έχετε περιφερειακή, πολυμερή, διαπεριφερειακή συνεργασία με τις χώρες ΑΣΕΑΝ, βλέπετε να απειλείτε αυτή η περιφερειακή συνεργασία ε, λόγω των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διμερώς με κάποια κράτη-μέλη της ΑΣΕΑΝ. Και μια τρίτη ερώτηση. Είχατε την καλοσύνη να πείτε δύο λόγια για τα νησιά Φίτζη και την Παπούα Νέα Γουινέα. Εδώ στο Κοινοβούλιο αξιολογήσαμε πολύ επικριτικά την κατάσταση στις νήσους Φίτζη ε, στην αξιολόγηση ενώ της εμπορικής μας οικονομικής συμφωνίας η σύνοψη της δικής μας συμφωνίας με τα νησιά Φίτζη Πώς νομίζετε ότι επηρεάζει ε, τις διαπραγματεύσεις για την επάνωδο στη δημοκρατία, της. καθυστερεί. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε να, να απαντήσω καταρχάς την τελευταία σας ερώτηση. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για μένα να εκφράσω άποψη για το αν ή ποια είναι η κατάσταση ε, θα επικρατήσει στο Φίτζι. Ε, μετά τα τελευταία γεγονότα. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, πιστεύω ότι Υπάρχει. Παρουσιάζεται μια ευκαιρία αρμονίας μεταξύ πολυμέρειας και διμερών ε, συμφωνιών. Η ε, αρμονία, ας πούμε η ισορροπία μεταξύ πολυμερών διαβουλεύσεων και διμερών είναι ένα θέμα κλειδί. Όπως πάντοτε δηλώναμε, η πολυμερής πτυχή και το εξειδικεύω αυτό ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης γιατί δεν συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί μου αλλά ε, ή μάλλον δεν πιστεύουν ότι ο ρόλος ε, των πολυμερών διαβουλεύσεων πρέπει να είναι πάντοτε στο ίδιο επίπεδο. Εγώ όμως πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουν παράλληλα και αρμονικά οι δύο αυτές, ε, τα δύο αυτά πλαίσια. Και απαντώντας την πρώτη σας ερώτηση. Ε, είχαμε δραστηριοποιηθεί έντονα στον πρώτο γύριο της Ντόχα, αλλά είχαμε μάλιστα δημιουργήσει την ομάδα του Κέρνς τότε και είχαμε προωθήσει ε, τα πρώτα συμπεράσματα του γύρου της Ουρουγουάης του αρχικού γύρου της Οριγουάης. Αλλά όπως ξέρετε οι εμπορικές ε, συμφωνίες δεν είναι ποτέ απλές διότι ο καθένας από τους συμμετέχοντες φέρνει τη δικιά του ατζέντα στο τραπέζι. Ακόμα και στις διμερείς διαβουλεύσεις για εμπορικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών υπάρχουν πάντοτε προϋποθέσεις, ε, κριτήρια ε, και συμφέροντα του καθενός που στο τέλος της ημέρας πολύ δύσκολα επιλύονται. Όμως θέλουν να πιστεύουμε ότι η Ντόχα δεν έχει πεθάνει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο τέλος της ημέρας και στο τέλος των προσπαθειών μας θα επικρατήσει η πολυμερής προσπάθεια. Διότι δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε το οικονομικό μέλλον αυτού του κόσμου σε διμερή βάση. Πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει την καθολική πτυχή, μια παγκόσμια πτυχή όλων των χωρών για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να είναι τα αποτελέσματα επικοδομητικά. Δεν έχουμε προκατηλημμένες απόψεις έναντι οποιασδήποτε οικονομικής μορφής, διακυβέρνησης και ακριβώς εκεί είναι και η δυσκολία της εξισορρόπησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια σωστή ισορροπία όμως, καμιά φορά τι να κάνουμε. Πρέπει να φροντίσουμε, παρόλες, παρόλο που δεν μας αρέσει, να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και εάν δεν είχα επιτύχει, αν δεν είχα αυτή την πολιτική βούληση, θα είχα παραιτηθεί από την πολιτική. Εγώ δεν είμαι μάγος, δεν έχω ένα μαγικό ραβδί που να μπορεί να διορθώνει τα λάθη. Αν είχα μαγικό ραβδί, θα είχα αποσυρθεί από την πολιτική και θα είχα ευχαριστηθεί τη ζωή μου. Ο... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Χόγκ, λέει ο πρέσβης, παρά την ιστορία και ιδιαίτερα τις παλινοδίες των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας προσπαθήσαμε να φέρουμε σε πέρα στον γύρο της Ντόχα. Ο Επίτροπος Ντεγκούχτ στάθηκαν σε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως όπως ξέρετε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Η ΙΠΑ, η Βραζιλία και η Ινδία γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες στον, κατά το τελευταίο μήνα, ιδιαίτερα στον ε, μη γεωργικό τομέα. Όπως είπε ο πρόεδρος Χόγκ, Προσπαθούμε να προωθήσουμε παράλληλα διμερείς συμφωνίες, επτά τέτοιες συμφωνίες προωθούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ε, τόνισε ότι θα ανοίξει τις αγορές της τομεακά, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ίση πρόσβαση από την άλλη πλευρά. Σε σχέση με τις νήσους Φίτζι και το οικονομικό πακέτο, Είμαστε πολύ ανήσυχοι από την αποτυχία της μεταβατικής κυβέρνησης, διότι δυστυχώς δεν τηρούνται οι δημοκρατικές αρχές. Αμείς μαζί με τη Νέα Ζηλανδία και άλλα έθνη είμαστε υπέρ των κυρώσεων ενώ επενδύουμε 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να ε, βοηθήσουμε τα νησιά Φίτζη μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βοηθά γενναιόδωρα τις χώρες του Ειρηνικού, είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, προσπάθησε να χορηγήσει αυτή την αρρωγή στα ε, νησιά Φίτζη για να προθεθεί αυτή η βοήθεια εμπρακτά. Και παράλληλα, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, μια συμφωνία πλαισίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας από τους τομείς ε, ε, σύναψη συμφωνιών αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης για ανθρωπιστική αρρωγή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα και στην Αφρικανική Ήπειρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρέσβη. Ο κύριος Ρόουτσεκ έχει το λόγο, που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνο για την Ασιατική Ήπειρο. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη νέα Ζηλανδία, διότι ο μεγαλύτερος εταίρος και ο πιο μακροχρόνιος είναι η Νέα Ζηλανδία ως προς εμπορικές συμφωνίες. Νομίζω ότι στο 1966 υπεγράφει η πρώτη συμφωνία. Μπορείτε να συγκρίνετε την ολοκλήρωση και όχι μόνο την οικονομική, γιατί μιλάμε και για ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Μπορείτε να συγκρίνετε την κατάσταση μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πού βλέπετε ομοιότητες και πού διαφορές. Το δεύτερο ε, ζήτημα είναι οι τριμερείς συμφωνίες, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, χώρες ΑΣΕΑΝ. Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που υπεγράφει τρία χρόνια πριν, από όσο γνωρίζω. Πώς εξελίσσεται. Γιατί οι χώρες ε, ε, ΑΣΕΑΝ αφορούν 400 εκατομμύρια καταναλωτών και είναι μια πολύ, μεγάλη, πολύ, πολύ μεγάλος χώρος για την Αυστραλία. Επίσης μιλήσατε και για διαπραγματεύσεις με την Κίνα και με την Ιαπωνία ως προς ε, σύναψη μιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει με αυτές τις χώρες και με αυτό το μπλοκ χωρών. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ως προς τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να σας δώσω έναν διεξοδικό κατάλογο διαφορών και ομοιοτήτων όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ μου και της Νέας Ζηλανδίας, γιατί δεν κατανοώ πλήρως τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση μεταξύ αυτών που ζείτε και γνωρίζετε εσείς και αυτών που γνωρίζουμε εμείς, αρκεί να πούμε ότι έχουμε κινηθεί πολύ κοντά ε, σε πολλούς τομείς μακροχρόνια ως προς ε, ένα ευρύ φάσμα όπως σας είπα ξεκινώντας από τα πρότυπα για τα τρόφιμα, τις προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Και ως προς την ελεύθερη διακίνηση μεταξύ χωρών υπάρχει ομοφωνία. η μόνη μεγάλη διαφορά, πέρα από αυτή που ήδη υπάρχει, είναι μια κοινοβουλευτική φύσης ένωση, η οποία δεν προβλέπεται στο εγγύς μέλλον, διότι υπάρχουν θέματα εθνικής κυριαρχίας και δεν ε, προσβλέπουμε σε αυτή την ανάγκη, δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη καθώς και θέμα κοινού νομίσματος μεταξύ μας. Κάτι τέτοιο δεν λήφθη υπόψη αρκετά σοβαρά. Συμμετείχα σε μία από τις έρευνες μιας κοινοβουλευτικής μας επιτροπής που ασχολήθηκε με ένα ευρύτερο ζήτημα, δηλαδή ένα κοινό νόμισμα στον νοτιοδυτικό ειρηνικό εξαιτίας του σχετικού πλεονεκτήματος των μικρότερων κρατών που έχουν εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Εάν είχαμε ένα κοινό νόμισμα, όπως το δικό σας ευρώ, και γνωρίζω βεβαίως ότι δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, όταν προτάθηκε κάτι τέτοιο δεν έτυχε ευρεία συνένεση στη δική μας περιοχή του κόσμου σε σχέση με τις συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες ΑΣΕΑΝ όπως είπε και ο πρέσβης χαιρόμαστε γιατί έχουμε ανοίξει τα εμπορικά μας σύνορα και μόνο έτσι θα αναπτυχθεί η οικονομία μας και το δεχόμαστε και από πλευράς Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Σε σχέση με τις ε, εμπορικές, ενδεχόμενες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, δεν γνωρίζω πώς εξελίσσεται το ζήτημα μέρα με τη μέρα. Γνωρίζω όμως ότι δεν θα συναυθεί μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κίνα στο εγγύς μέλλον. Δεν είναι καθόλου απλή η διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ως προς τις σχέσεις μας με την Κίνα. Απλώς έχουν ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης του επιχειρήν και επειδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων και εμείς θα θέταμε ένα περιορισμένο αριθμό θεμάτων επιτάπητος, ε, το ζήτημα θα, είχε, θα μπορούσε να έχει διαφορετική εξέλιξη. Ως προς την Ιαπωνία θα προτιμούσα να μην σχολιάσω. Ο πρέσβης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι η Κίνα ε, είναι ο πρώτος εμπορικός μας εταίρος. Ήταν ο δεύτερος ε, μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την οικονομική κρίση Κυρίως σε θέματα ε, παιδείας έχουμε συνεργασία και ανταλλαγές, ε, αλλά και σε εμπορεύματα στον άνθρακα. Ο Πρωθυπουργό μας θα επισκεφθεί την Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει. Είναι ο τρίτος εμπορικός μας εταίρος η Ιαπωνία. Και σε σχέση ε, με την ΑΣΕΑΝ και τη, τις ελεύθερες, ε, συναλλαγές ελεύθερου εμπορίου, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Είναι πραγματικά πάρα πολλέ Έχουν μια πληθώρα συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες της ΑΣΕΑΝ. Αλλά δεν συνιστά αυτό καμιά ειδική απειλή για τις σχέσεις μας με τις ε, χώρες του ΑΣΕΑΝ. Αφήστε δε που και να ήταν απειλή θα την εθαρρύναμε να συνεχίσει προς την κατάσταση, ε, την κατεύθυνση αυτή. Εμείς Δεν επιθυμούμε τέτοιου συμφωνία. Η βασική μας δέσμευση είναι η πολυμερής ε, ε, συνεργασία στα πλαίσια του ΠΟΕ που γνωρίζετε ότι αγωνιζόμαστε εκεί. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, και άλλες παρεμβάσεις. Έχουμε μισή ώρα μπροστά μας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούμε δύο ομιλητές και μετά να σας δίνουμε τη δυνατότητα να απαντήσετε κύριε Πρόεδρε για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Καζάκ, μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε ε, Πρόεδρε Χόγκ, Αγαπητοί συνάδελφοι, με ζωηρό ενδιαφέρον άκουσα την παρουσίασή σας σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων του γύρου της Ντόχα και τις σχέσεις με την ε, Αυστραλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό μας ενδιαφέρει πολύ η έκβαση για να δώσουμε και μια νέα όθηση ακριβώς στην πολυμερή ε, συνεργασία ε, και στον εμπορικό τομέα και όχι στις διμερείς συμφωνίες. Αναφερθήκατε ακριβώς σε διμερείς συμφωνίες που έχετε εσείς με την Κίνα και την Ιαπωνία. Θα ήθελα όμως να σας κάνω μια ερώτηση γιατί διάβασα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία προς την κατεύθυνση αυτή θα ξεκινήσουν φέτος. Ίσως γνωρίζετε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνάψει τέτοιου είδους συμφωνία με την Ινδία, αλλά έχουμε δυσκολίες κυρίως από ινδικής πλευράς με τις ρήτρε αηφόρου ανάπτυξης και ε, κάποιες ε, άλλες ρήτρε που αφορούν την παιδική εργασία και άλλα ατινά. Εσείς τι πιστεύετε θα μπορούσατε να συναντήσετε εμπόδια στη με την Ινδία για αυτό το θέμα. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Το διμερές εμπόριο Αυστραλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε ανητικό ισοζύγιο για την Αυστραλία. Οι εισαγωγές σας είναι τριπλάσιες από τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς προτίθεστε να αντιστρέψετε αυτή την τάση, να την ξεπεράσετε και να επέλθει μεγαλύτερη ισορροπία στις διμερείς μας σχέσεις. Ευχαριστώ κύριο Σίβιτς. Ευχαριστώ. Προέρχεστε από μια ε, περιφέρεια του κόσμου η οποία απέχει πάρα πολύ από την Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεσπόζει η Κίνα από εκείνο το μέρος του κόσμου. Μιλάμε για την οικονομική σημασία της Κίνας. Είναι μια αναδυόμενη χώρα. Ποια είναι η προοπτική της Αυστραλίας, ε, ποιες είναι οι προοπτικές ως προς τις σχέσεις σας με την Κίνα Ποια είναι η άποψή σας μεταξύ διαλόγου Κίνας και Ταϊβάν μέσα στα πλαίσια της ενδεχόμενης ενοποίησης των δύο χωρών. Έχετε το λόγο αν θέλετε να απαντήσετε και στους δύο συναδέλφους. Έχετε το λόγο. Καταρχάς, η ερώτηση για τις διαπραγματεύσεις με την Ινδία. Εμείς βέβαια δεν θα παραλείψουμε ε, να επισημάνουμε προβλήματα όπως η παιδική εργασία ή κάτι το οποίο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τονίζει την έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως αυτό επαφίεται στους διαπραγματευτές. Εγώ δεν ε, παρακολουθώ από κοντά τις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι βέβαιος ε, ότι θα εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου είναι αποδεκτή και συμβατή με τα κανονικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδεκτή από το λαό μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι μας θεωρούν ε, ε, αξιόπιστους και ότι έχουν εμπιστοσύνη σε εμά. Εάν είχα ο ίδιος συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις θα, θα είχα περισσότερες προφορίες, αλλά δεν έχω. Όσον αφορά το έλλειμμα που μπορεί να υπάρχει μεταξύ μας στις εμπορικές συναλλαγές, εμείς δεν το θεωρούμε αυτό ε, απαραίτητα ως θέμα, τη πρόβλημα ελευθέρων συναλλαγών, των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Αλλά πολλές φορές στις εμπορικές συναλλαγές και στις υπηρεσίες, σε έρευνες, σε εκθέσεις τις οποίες έχω δει από το παρελθόν, διαπίστωση υπάρχουν πάρα πολλά προσκόμματα, ιδίως ε, δασμολογικά. Έχουμε Έχουμε ε, σχετική εμπειρία, ιδίω σε χρηματοοικονομικά θέματα και επίσης τα θέματα του τουρισμού, της παιδείας και ε, εκεί, σε αυτούς τους τομείς, ορισμένα τεχνητά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν για να ανθίσει περισσότερο η συνεργασία. Επίσης η αγροτική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική για μας. Από τη στιγμή που εμείς έχουμε τεράστια αποθέματα φυσικών πρώτων υλών ε, που μπορούμε να εξαγάγουμε και που δεν υφίστανται δασμολογικές ε, ε, δασμολογικά προσκόμματα, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε αυτές τις εμπορικές συναλλαγές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η απάλληψη δασμολογικών εμποδίων ανοίγει τεράστιες, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Όσον αφορά τώρα την κυρίαρχη θέση της Κίνας, τα τελευταία 30 και χρόνια είχαμε μία θα έλεγα καινοτομική προσέγγιση προς την Κίνα όταν δεν ήταν της μόδας οι σχέσεις με την Κίνα ή δεν ήταν δυνατό να υπάρχουν και ε, διαδοχικές κυβερνήσεις διαφορετικών αποχρώσεων βελτίωσαν και ανέπτυξαν αυτές τις σχέσεις. Πιστεύουμε ότι η Κίνα είναι ένας βασικότατος παίκτη στο μέρος αυτό του κόσμου και πρέπει να συμμετάσχουν δραστήρια στις, στη συνεργασία μας, στο διάλογο, στις διαβουλεύσεις, για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα Κίνας-Ταϊβάν, αυτό άπτεται ε, του, του, όλου θέματος της σταθερότητας της περιοχής. Έχουμε εδώ και ε, πολύ καιρό υιοθετήσει μία συμφωνία ότι υπάρχει μόνο μία Κίνα, μία Κίνα, μία είναι η Κίνα και πάντοτε λέγαμε ότι αναγνωρίζουμε μία μοναδική Κίνα και για την Ταϊβάν λέγαμε πάντοτε ότι είναι μία οικονομική οντότητα. Οι Κινέζοι έχουν κατανοήσει απολύτως τη θέση μας και βεβαίως καλωσορίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταξύ των δύο οικονομιών να συγκεράσουν τις προσπάθειές τους υπό μία οντότητα και να αναγνωρίζονται ως μία οικονομική και διπλωματική οντότητα. Αυτές οι προσπάθειες βέβαια δεν μας έχουν εμποδίσει όπως ε, καταλαβαίνετε να υποστηρίζουμε τα πρώτα βήματα του IPEC, δηλαδή της, ε, ε, του πλαισίου συνεργασίας Αυστραλίας ε, και Ειρηνικού. Αυτό το πλαίσιο συνεργασίας του APEC έχει λειτουργήσει πολύ σωστά, πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και η Κινέζικη κυβέρνηση έχει σεβαστεί την προσέγγιση μας η οποία επαναλαμβάνω λέει ότι η πολιτική μας ε, αφορά μία Κίνα και μόνο μία. Ο πρόεδρος. Ο Ρόμπερτ Στέρντι έχει το λόγο που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν. Καταρχήν, αυτό έχουμε τον κύριο ε, Hans Pöttering στο ακροτήριό μας Um, Πρώτη φορά που το συνάντησα δεν είχαμε ούτε μία άσπρη τρίχα στο κεφάλι μας. Αυτό είναι πολλά χρόνια πριν. Και ο κύριος Πέτερινγκ έσυξε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα ε, και τις συζητήσεις που έχουμε στο ερχόμενη Κυριακή ε, το γεγονός ότι έχουμε μία ειρηνική, την εγγύηση μιας ε, ειρήνης και μιας ειρηνικής ζωής στην Ευρώπη είναι τόσο σημαντικό την Κυριακή θα γιορτάσουμε λοιπόν ε, αυτή την ειρηνική περίοδο και εσείς ήσασταν ένας από τους προτεργάτες της επιτυχίας της. Εγώ είχα εργαστεί τότε υπό τον γύρο της Ιρουάης και πιστεύετε ότι ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσει να αποτελεί, προβλήματα, ε, να αποτελεί πρόβλημα βλέπουμε τις τεράστιες αυξήσεις των τιμών των, της των σιτηρών πάνω από 200 δολάρια ο τόνος τι θα γίνει με την πολιτική της ελευθερίας της αγοράς έχουν ανέβει ε, εξουθενωτικά οι τιμές ε, και με την, τον αυξανόμενο πληθυσμό είναι απίστευτο. απίστευτος ο όγκος των τροφίμων που χρειάζονται για τη διατροφή ε, ε, παγκόσμια του πληθυσμού. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα η αύξηση αυτή, η αλματώδης αύξηση των τιμών. Πώς το αντιμετωπίζετε. Επίσης, αυτό που πρόσεξα στο briefing και επειδή αυτή είναι μια κοινή συνεδρίαση με τις εξωτερικές ε, υποθέσεις είπατε ότι η, Αυστρα... κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει επιβεβαιώσει την πολιτική της δέσμευση ανακοινώνοντας τον Απρίλιο του 2011 μία νέα εμπορική πολιτική. Και είπατε ότι αυτή η εμπορική πολιτική θα αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τις επιπλοκές ε, ή από τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι τελείως αντίθετο με αυτά τα οποία συζητάμε εδώ, τη διασύνδεση εμπορίου και πολιτικής. Ο κύριος Ντανζάν, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας, που θα αναφερθεί φαντάζομαι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για το τι ζήσατε στο Queensland φέτος το χειμώνα. Εγώ επισκέφτηκα την Καλιδονία και γνωρίζω το μέγεθος των καταστροφών που γνωρίζετε και εσείς. Βεβαίω μιλάμε για μεγάλη οικονομική ε, δέσμευση όλων των κρατών σε αυτό το τομέα. Ποια είναι η δική σας ε, πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν, ε, υπάρχει κατάσταση δημοσιονομικής λιτότητας σε σχέση με τις ε, αμυντικές σας δαπάνες. Επίσης, σε σχέση με την ε, κοινή αμυντική πολιτική και την εταιρική μας σχέση με την Αυστραλία, επειδή υπάρχουν κοινέ στρατιωτικές ασκήσεις και επειδή έχουμε μια κοινή ναυτική δύναμη που καταπολεμά την ε, πειρατεία στη Σομαλία, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα state building στον ε, τομέα της δικαιοσύνης, των ε, τελωνιακών αρχών και ούτω καθεξής. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε σαστε να είσαστε πραγματικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο είναι ευκταίο. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, σε σχέση με το θέμα των εμπορικών ε, σχέσεων. Εγώ εδώ και ε, τρεις εβδομάδες ταξιδεύω, άρα δεν το γνωρίζω. Δεν ε, πρόκειται για το γεγονός ότι η κυβέρνησή μου δεν μου λέει τίποτα, αλλά εγώ βρίσκομαι καθοδόν και σε επισκέψεις ανά τον κόσμο. Ίσως ο πρέσβης γνωρίζει την κατάσταση, όμως Δεν μπορεί κανείς να απομακρυνθεί, να μην λάβει υπόψη τον ε, τομέα της ε, γεωργίας. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των μελημάτων μας. Και ε, άκουσα την δήλωσή σας. Δεν ξέρω κατά πόσο οι δυνάμεις αγοράς θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν από μόνες τους. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται κάποια μορφή παρέμβασης. Και ως προς την ε, δήλωση περοεμπορικών ε, σχέσεων υπουργικού επίπεδου, θα αφήσω τον ε, πρέσβη να σας απαντήσει. Ως προς τις αμυντικές δαπάνες, ανταποκρινόμαστε στις δεσμεύσεις μας. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καθοδική πορεία δαπανών. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα ψηφιστεί στις 12 Μαΐου, θα υποβληθεί από την κυβέρνηση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι πρωτοβουλίες θα ληφθούν από πλευράς κυβέρνησης. Δεν το γνωρίζω μέχρι τώρα, αλλά θα με εξέπλητε εάν μειώνονταν οι αμυντικές μας δαπάνες. Εμείς είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και δραστήριοι, όπως γνωρίζετε, και στο Αφγανιστάν έχουμε σοβαρές δεσμεύσεις, σοβαρή δέσμευση και στην ειρήνευση αυτής της περιφέρειας και ενώ δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, συμμετέχουμε στις ασκήσεις έτσι ώστε οι δυνάμεις μας να χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις, ε, στην κοινή αυτή δύναμη. Βεβαίως ως προς τη Λιβύη βρισκόμαστε πολύ μακριά και δεν θα είχαμε τα κατάλληλα μέσα. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ραντ, διαδραμάτισε θετικό ρόλο για την εφαρμογή της ζώνης ε, μη πτήσεων. Ως προς τη στρατιωτική μας δέσμευση, από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, Εξωτερικών θεωρούμε ότι διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο. και τη στιγμή που υπάρχει μία σύραξη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά την ανακοχή στην Κύπρο, αν μπορώ να μιλήσω για ανακοχή, οι ομόσπονδες αστυνομικές δυνάμεις βοήθησαν και δεν έχουμε φυστεί μέσον προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς θέματα πειρατείας και ούτω καθεξής, θα μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα μέσα στα πλαίσια του θεάτρου επιχειρήσεων. Και υπάρχουν μέσα αντιμετώπισης ε, της ε, παράνομης ε, μετανάστευσης και αυτό το αντιμετωπίζουμε και με την ακτοπλοεία μας, τις ακτοπλοϊκές δυνάμεις και τις τελωνιακές αρχές. Επίσης, υπάρχει εξοπλισμός μέσα στα πλαίσια και των επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως ε, περιπολούμε και τις ακτές μας έτσι ώστε να ανταποκριθούμε ως προς τις αμυντικές μας δαπάνες και δαπάνες ασφαλείας για να προωθήσουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις την ειρήνη ανά τον κόσμο. Και ο πρέσβης θα με συμπληρώσει στα θέματα που δεν απάντησα. Σας ευχαριστώ. Ακούτε τον πρώην Υπουργό Αμήνης της Αυστραλίας. 2% μόλις του προϋπολογισμού είναι αμυντικές δαπάνες και την τελευταία δεκαετία εξυγχρονίζουμε η σημερινή κυβέρνηση. Έχει δεσμευτεί για το 3% ε, πραγματική ετήσια αύξηση των αμυντικών δαπανών την επόμενη δεκαετία. Ταυτόχρονα όμως να πιάνουν τόπο τα χρήματα αυτά στις αμυντικές δαπάνες. θεωρούμε ότι η ασφάλειά μας ε, βασίζεται και ε, σε συμμαχίες, όχι μόνο στην περιοχή και γύρω από τα σύνορά μας, αλλά και παγκόσμια. Με το ΝΑΤΟ, ας πούμε, διαπραγματευόμαστε μια στρατηγική συνεργασία για την αντιμετώπιση της πειρατείας, την αντιτρομοκρατία και ε, βοήθεια σε περίπτωση θεομηνιών και όχι μόνο με το ΝΑΤΟ αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεργαζόμαστε παγκοσμίω, γιατί έχει μια παγκόσμια αντίληψη για τα θέματα ασφαλείας και όπως είπε και ο, ο Πρόεδρος είμαστε ε, η δέκατη ε, συμμετοχή κατά σειρά, ε, κατά μέγεθος ε, στο Αφγανιστάν, περισσότερο από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ. Επίσης ενεργά συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση της πειρατείας ε, και τέτοια ζητήματα. Τώρα σε σχέση με το εμπόριο, την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ουσιαστικά αλλά στάση στις διαπραγματεύσεις, στις εμπορικές. Βεβαίως, συνεχίζουμε να ανησυχούμε για θέματα όπως είναι η παιδική εργασία, ή καταχρήσεις, ε, εκμετάλλευση εργαζομένων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά η Ινδία ε, μάλλον ε, εμείς έχουμε δηλώσει ότι θα ανοίξουμε τις αγορές μας ακόμα και αν κάποιοι άλλοι δεν τις ανοίξουν συνομιλητές. Και επίσης δεν θα είναι διακοσμητικού χαρακτήρα η διαπραγματεύση ανακοίνωση κυβέρνηση, αλλά θα είναι ουσιαστικές. Και επίσης ήθελα να τονίσω ότι παρόλο που έχουμε 40% του ε, ε, παγκόσμιου επιφανειακού ουρανίου, δεν θα πουλήσουμε ουράνιο στην Ινδία γιατί δεν έχει ε, προσχωρήσει στη συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο οικονομικά συμφέροντα αλλά και αρχές. Και ακριβώς επειδή σήμερα βρισκόμαστε σε ισχυρή οικονομική θέση, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή τα τελευταία 40 χρόνια ανοίξαμε τι αγορές μας παντού και κάναμε και μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό είμαστε σημερινή ισχυρή θέση. Και αποφάσισε η κυβέρνηση ότι είναι προ το δικό μα συμφέρον να ανοίξουμε τις αγορές μας ε, για μεγαλύτερη ευημερία. Ευχαριστώ. Ε, ε, ο κύριος Κύριλοβ και ο κύριος Γεωργίου και μετά κλείνει η συζήτηση. Λόφ. Κύριε Κερουσιαστά, αναφερθήκατε στην δέσμευσή σας και την εμπλοκή σας στο Αφγανιστάν. Ε, προφανώς θα γίνονται ορισμένε συζητήσεις στην Αυστραλία για το αν είσαστε αποτελεσματικοί ε, εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο πώς αξιολογείτε τη γενική κατάσταση στο Αφγανιστάν και την ενδεχόμενη στρατηγική εξόδου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Θέλω να ακολουθήσω και εγώ τον κύριο Χοκ. Ε, άκουσα την περιγραφή σας για την οικονομία της Αυστραλίας και χάρηκα γι' αυτό γιατί την περιγράψατε με πολύ θετικά λόγια. Να μου επιτρέψετε να πω ότι μου θύμισε λίγο τις ε, θετικές αναφορές και αναλύσεις που γίνονταν στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής μόνο 10 δευτερόλεπτα πριν την εκτόξευση αυτής της μεγάλης παγκόσμιας κρίσης. Ε, δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις βέβαια, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι διαφορετικό κάνετε εσείς στην Αυστραλία που μπορούσε να αποτελέσει και παράδειγμα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για μας. Για το μεταναστευτικό είπατε ότι σας προβληματίζει και ότι αντιμετωπίζετε, έχετε κι εσείς αυτό το μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε. Ε, αφήνοντας πίσω τελείως, αν μου επιτρέπετε, την διπλωματική γλώσσα, εγώ νομίζω ότι το αντιμετωπίζετε. Η χώρα των πρώην μεταναστών, που είναι η Αυστραλία, αντιμετωπίζει τους νυν μετανάστες με χιλιάδες διαδηλωτές πρώην μετανάστες στα παράλια να αντιστέκονται μέχρι τελικής πτώσεως στο να μην μπουν στη χώρα καινούργιοι μετανάστες. Το τρίτο το έχει βάλει ο κύριος Κυριλόφ πριν από λίγο που αφορά το Αφγανιστάν. Θα ήθελα την πρόβλεψή σας για το μέλλον, μέχρι πού θα πάει η παρουσία σας εκεί και τι προβλέπετε. Ευχαριστώ. Eh, Ο πρόεδρος Γερουσίας ε, έχει το λόγο για τα συμπεράσματά του. Καταρχήν ως προς το Αφγανιστάν, Εμείς συμμετείχαμε με βάση την απόφαση της κυβέρνησης και όχι απόφαση του Κοινοβουλίου. Όμως, φέτος δαπανίσαμε αρκετό χρόνο και στην Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να συζητήσουμε τα υπέρ της συμμετοχής μας στις στρατιωτικές δυνάμεις του Αφγανιστάν. Και αν και υπήρξαν ε, ορισμένες ε, αμφιβολίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα δεν υπήρχε ευρεία υποστήριξη για τη συμμετοχή μας στο Αφγανιστάν. Ίσως άλλοι θα επιθυμούσαν κάτι διαφορετικό προς τη λήψη της απόφασης, τον τρόπο λήψης της απόφασης, αλλά υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος, όχι την παρουσία μας. Ως προς μια στρατηγική εξόδου, εμείς ε, έχουμε αποστείλει ειδικέ δυνάμεις, ειδικέ στρατιωτικές δυνάμεις, και επίσης ε, ειρηνευτικές δυνάμεις, δυνάμεις ανοικοδόμησης της χώρας, γιατί θεωρούμε ότι μία εμπόλεμη κατάσταση δεν αρκεί, ούτε θα είναι επικερδής. Γι' αυτό έχουμε αποστείλει μηχανικούς και άλλους που βοηθούν τους Αφγανούς για την ε, ανοικοδόμηση της χώρας για να χτίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου να ζήσουν και να υπάρχει αξιοπρέπεια και προώθηση της αυταξίας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Βεβαίως γνωρίσαμε απώλειες, όπως είναι γνωστό, στο Αφγανιστάν και αυτή η απώλεια ήταν πολύ μεγάλο τίμημα που πλήρωσαν πολλές οικογένειες της Αυστραλίας. Είτε ε, είμαστε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε στη Γερουσία αποτίσαμε μεγάλο φόρο τιμής για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ε, ανά τον κόσμο. Και αυτό ξεκινά από την ε, Καλή Πολύ όπου θα ε, μεταβούμε για, την, για να γιορτάσουμε την επέμβαση και των δυνάμεων της Αυστραλίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Συμμετείχαμε και εκεί. Πάντα ήμασταν ένα έθνος που είχε ταχθεί υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης ανά τον κόσμο. Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση της οικονομίας και τα θετικά σχόλια που έκανα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αντίτιμο και στη δική μας οικονομία και θα συμφωνήσει και ο πρέσβης μαζί μου. Δεν μιλάμε για ε, μια πλήρη επιτυχία και απόλυτη επιτυχία και ελπίζω να μην καταρρεύσει η οικονομία τις επόμενες ημέρες επειδή εγώ την υπερασπίζομαι τόσο στεναρά. Πιστεύω σε σχέση με τις είπα και ό,τι αντιμετώπισαν άλλες χώρες ως προς την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εμείς προβάλλουμε μια υψηλή ρύθμιση η οποία δεν θα επέτρεπε να συμβούν αυτά που συνέβησαν στην αγορά των ΙΠΑ και άλλες αγορές. Και εάν δείτε τι συνέβη σε επίπεδο G20 σε σχέση με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, θα δείτε ότι η Αυστραλία τάχθηκε υπέρ της μεγαλύτερης ε, οικονομικής, των μεγαλύτερων δεσμεύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Δηλαδή δεν είμαστε υπέρ της ελεύθερης ρύθμισης των ε, δυνάμεων της αγοράς, της αυτορύθμισης, γιατί έτσι λειτουργήσε η αγορά των ΗΠΑ και αυτό οδήγησε στη, στον όλεθρό της Εάν εξετάσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδιαίτερα τις δικές μας, προσπαθούμε να τις ε, ρυθμίσουμε. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ε, λογοδοσία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παράνομες δυνάμεις οι οποίες δρούν κατά του κανονιστικού αυτού πλαισίου. Ως προς τη μετανάστευση, θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε δύο ζητήματα. Τους παράνομους μετανάστες που παραμένουν παραπάνω στη χώρα με το σύστημα των θεωρήσεων έρχονται με τουριστική βίζα και μένουν παραπάνω από όσο τους επιτρέπει η θεώρηση. Υπάρχουν 60.000 παράνομοι μετανάστες οποιαδήποτε χρονική στιγμή που σε αναλογία με το ε, πρόβλημα σε άλλα μέρη της Ευρώπης είναι αμεληταίο. Ως προς εκείνους που διαλέγουν το πιο επικίνδυνο δρόμο, να προσέθουν δηλαδή διαφαλάσεις έχουμε άμεση υποχρέωση να ακολουθήσουμε τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών είτε αποζητούν άσυλο είτε δεν υπησέρχονται σε αυτή την κατηγορία. και δεν τους χορηγείται άσυλο, άρα δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Βεβαίως γνωρίσαμε τέτοια μεταναστευτικά κύματα. Και έχουμε τις ε, κατάλληλες, διευρύναμε τις υποδομές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εντάχει πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αιτήματα χορήγησης ασύλου. Έχουμε υποχρεώσεις και πολλοί βεβαίως κρατούνται. Αυτό όμως δεν γίνεται σε γυναίκες και παιδιά. Αυτή είναι η κυβερνητική μας πολιτική. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Πού θα οδηγήσουν όλα αυτά δεν το ξέρω. Πολλοί παράνομοι μετανάστες προέρχονται από το Αφγανιστάν, άλλοι από τη Σρι Λάνκα και από αλλού όπως το Ιράν. Αλλά οι ροές είναι εποχικού χαρακτήρα στην ε, περίοδο μουσώνων είναι πολύ δύσκολο να έρθουν διαθαλάσσεις ε, στα βορειοδυτικά της Αυστραλίας. Και έτσι υπάρχει μια επιβράδυνση προσελεύσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέσβης θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Μετά από 40 χρόνια μεταρρύθμισης πολιτικής υφής και κυβερνητικής αντιμετωπίσαμε το, το θέμα των μεταναστών. Εμείς είμαστε ένας υπερήφανος λαός μεταναστών και έχουμε πολύ μικρό και αμεληταίο πρόβλημα μετανάστευσης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως ο συνάδελφος Στέρντι θα ήθελε να χαιρετήσει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να ευχαριστήσω τον γερουσιαστή και τον κύριο Πρέσβη για τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις τους σε πάρα πολύ διαφορετικά θέματα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ε, παρακολουθούμε βεβαίως και τα αθλητικά ε, συμβαίνοντα στην Αυστρία και το κρίκετ και σε άλλα σπορ. Εκ μέρους της Επιτροπής σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Συμφωνούμε όλοι βεβαίως και σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε εδώ μεταξύ μας. Good to see you. Good to see you. Ωραία, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο με, με, με θέμα της ημερησίας διάταξης. Είναι η έκθεση της κυρίας Μουνίτ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο φορέα στα πλαίσια των πολυμερών οργανώσεων. 154 ε, είναι οι τροπολογίες και η συγγήτρια έχει συντάξει 10 τροπολογίες συμβιβασμού. Ευχαριστώ. Η παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή η συλλογική διαχείριση των κοινών προβλημάτων μας, γνωρίζει μια κρίσιμη συγκυρία, γιατί έχουν αυξηθεί γεωμετρικά τα θέματα της διεθνούς ατζέντα και σε περιπλοκότητα και σε αριθμό και έχουμε ε, διεθνείς οργανισμούς και κράτη που βρίσκονται στα όρια πλέον των δυνατοτήτων διαχείρισης. Συζητούμε τώρα τη μεταρρύθμιση των διεθνών οργανισμών που έχουν σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ε, συζητούμε για το πώς θα τις προσαρμόσουμε αυτές τις οργανώσεις στη νέα διεθνή πραγματικότητα. Αφενός για να ανταποκριθούμε στις αδυναμίες των διεθνών οργανισμών που είναι απαρχαιωμένες ας πούμε γιατί από την άλλη πολλαπλασιάζονται οι άτυπες ομάδες, κλαμπ, λέσχες, ενώσεις και τα λοιπά για να ασχοληθούν με ειδικά θέματα της διεθνούς ατζέντα. Θα πρέπει να δούμε τι νομιμότητα έχουν αυτές οι νέες οντότητες και τι συνοχή και να καθορίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός αυτών. Από την άλλη ο πολυ ε, πολικός κόσμος μας δυσκολεύει τη διεθνή διακυβέρνηση γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει παγκόσμιο στρατιωτικό πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ άλλων έχουν πρόβλημα με τις εσωτερικές δομές της. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει πώς ε, συντονίζεται με τα άλλα κράτη-μέλη στους παλιούς και νέους οργανισμούς. Αυτά ε, σε γενικές γραμμές είναι το πλαίσιο το οποίο συζητούμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο. 154 τροπολογίε κατατέθηκαν. Καταφέραμε να φτάσουμε σε 10 συμβιβαστικέ που ομαδοποιούν 52 από τις τροπολογίε αυτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου, καθόλου σεβαστές και αποδεκτές οι υπόλοιπε τροπολογίε που δεν έχουν μπει στου συμβιβασμού. Απλώς δεν μπορούσαν να ενταχθούν από το αντικείμενό του. Γιατί θεματικά απήχαν Οπότε χρειάστηκαν ξεχωριστές παραγράφους. Λοιπόν, η έκθεση αυτή με τις δικές σας τροπολογίες νομίζω μπορεί να είναι συνενετική σε γενικές γραμμές στην Επιτροπή μας, διότι δεν είναι πολιτικής φύσεως, είναι μάλλον θεσμικής, θα το χαρακτήριζα ε, το θέμα. Ποιοι είναι οι οργανισμοί, ποιες δυνατότητες και μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα μεταρρυθμίσει και πώς μπορεί με τα νέα μέσα βασικά που είναι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, που τα θέτει ε, σε στη διάθεση της Ένωσης πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε διεθνώς. Ίσως η μεγαλύτερη πολιτική διαφορά μεταξύ των πολιτικών ομάδων να είναι το θάρρος και το σθένος με το οποίο θα αντικαταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη της, ιδιαίτερα εκεί που έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες η Ένωση και πώς θα συντονίζεται για να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη στους διεθνείς οργανισμούς. Και πώς θα εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και πώς θα συνεργάζεται μαζί τους εκεί που έχουν οι συντρέχουσες αρμοδιότητες. Αυτές είναι λοιπόν οι συμβαστικές τροπολογίες. Να σας εξηγήσω εν συντομία Συμβαστική υπαριθμών 1 ομιλεί για την ανάγκη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, ενεργειακή ασφάλεια, καταπολέμηση ένδυση, κλιματική αλλαγή, καταπολέμηση ε, ε, της παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη ε, συμβαστική τροπολογία, ποια είναι η διεθνής προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς έχει συμμετοχή της Είπα τι εκπρόσωπος επίσης τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και πώς εξασφαλίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή και εκεί που έχει επαναλαμβάνω αποκλειστικές αρμοδιότητες και εκεί που έχει συντρέχουσες αρμοδιότητες και τις μοιράζεται με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι ενιαίο το μήνυμά μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και στα κράτη-μέλη, εκεί που διατηρούν την αντιπροσωπεία τους. Τρίτη τροπολογία. Σήμερα η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς είναι ε, συγκεχημένη, κατακαιρματισμένη και ad hoc. Χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό για να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερο το δυναμικό τη συνθήκη Λισαβόνα και να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερεί οργανισμού. Συμβαστική υπαριθμών 4. Αναφέρεται κυρίω στους πολυμερείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εξηγούμε γιατί οι δημογραφικές αλλαγές εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάσσουν ανακατανομή των θέσεων και τη στάθμιση των ψήφων στους πολυμερείς οργανισμούς και ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει τη δυνατότητα όσο και την προθυμία ε, αλλαγής και προσαρμογή στι σημερινέ συνθήκες, δηλαδή στο εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για παράδειγμα, ζητούμε ε, ε, συνεργασία για την αηφόρο ανάπτυξη, για την ε, κρίζωσή της ένδυας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής. Συμβαστική παριθμό 5. Παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερεθνικού φορέα με περιφερειακό χαρακτήρα, της οποίας η νομιμότητα απορρέει από συνθήκες επιτρέπει να στήσει ένα διεθνές όργανο βελτιωμένο σύμφωνα με ε, την ατζέντα μας και με τις αρχές και τις αξίες μας. Αν θέλει να είναι παγκόσμιος πρωταγωνιστής χρειάζεται να ε, είναι καλύτερος ο συντονισμός και διεθνώς και να ακούγεται με μία φωνή προς τα έξω. Αυτό είναι εκ των όνου κάνευ για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ιδιαίτερα την ανάγκη να ενισχυθεί η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας ή της ε, προστασίας και της ευθύνης που έχουμε να προστατεύουμε τον πληθυσμό και ε, θα συμπεριλάβουμε ε, αυτή την ιδέα. Έκτη συμβαστική τροπολογία είπα ότι εκπρόσωπο συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσουν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια διακυβέρνηση και να δουν ποιες είναι οι δυνατότητες ε, υλοποίησης αυτών σε συνεργασία πάντα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έβδομη, τι γίνεται σε περίπτωση Ε, άσκηση καθηκόντων σε τομεί που η Ένωση έχει αποκλειστικέ αρμοδιότητες. Καλούνται τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στους οργανισμούς αυτούς. Μήπω θα πρέπει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί να εκπροσωπεί και τα 27 κράτη-μέλη. Και εν πάση περιπτώσει να στηρίξουν τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν δεν παρετούνται από τη συμμετοχή του στον οργανισμό αυτό. Παράδειγμα, ο ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστικέ αρμοδιότητε εκεί και ηγείται τη θέση στον ΠΟΕ σε ε, ό,τι αφορά τις συντρέχουσες αρμοδιότητες. Ο κανόνας θα πρέπει να είναι συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αλλά με κάποιο πρώτερο συντονισμό. Στην έκθεση, σε κάποια συμβαστική τροπολογία, γίνεται λόγος για αναζήτηση μια θέση προηγούμενου συντονισμού, δηλαδή των κρατών μελών, για να μην πέφτουμε σε αντιφάσεις όσο γίνεται και να μην ακούγεται μια κακοφωνία προς τα έξω, γιατί θα είναι και οπισθοδρόμηση. Και όπου υπάρχει ε, διχογνωμία, ανταγωνισμός τη εκπροσώπηση να κάνουν ένα βήμα πίσω τα κράτη-μέλη, να υποχωρούν μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούγεται εκείνη προ τα έξω και να φαίνεται. Σε αυτό αναφερόμουν όταν έλεγα ότι η μόνη διαφορά είναι σε ποιο επίπεδο δημοκρατίας θέλουμε να εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαστική παριθμών 8 αναφέρεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στηρίζουμε, όπως επανειλημμένα έχει πει σε εκθέσεις του Κοινοβούλιο, μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προτείνεται προοδευτική αντικατάσταση του δικαιώματος ε, βέτο, ε, ένα σύστημα υπερενισχυμένης πλειοψηφίας και επίση φιλοδοξεί μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ζητούμε από την ύπατη εκπρόσωπο ως ε, προεδρεύουσα του Συμβουλίου Εξωτερικών να ε, κάνει τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εκπροσωπούν τις θέσεις του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαστική 9 ε, αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ είχε κάνει πολλέ τροπολογίε η κυρία Ανδρικά ε, γίνεται λόγος για το ποιο είναι μέλος εκεί για να αποτραπεί ε, το φαινόμενο χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχουν έδρα εκεί. Επίσης ζητείται να συσταθεί η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατία στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις αντιπροσωπείες ε, του Συμβουλίου και Επιτροπής στη Γενέβη να συσταθούν το συντομότερο δυνατό. Και τελευταία συμβιβαστική υπαριθμών 10 αναφέρεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης επειδή ε, προσχωρεί στην ΕΣΔΑ, τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούμε να μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα των 10 συμβαστικών τροπολογιών και νομίζω ότι καταρχήν δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις πολιτικές ομάδες γιατί συνεννοηθήκαμε τους κοιόδης ηγητές και τα συνενώσαμε. Ευχαριστώ τον Πίτερ Βάχτα και την ε, Γραμματεία για τη πολύτιμη βοήθεια του και μαζί με τους κοιόδης ηγητές. Ε, Ωραία, συνεχίζουμε με τους σκιώδεις. Ο κύριο Κούκαν έχει το λόγο πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για την εργασία της ε, επί της και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για τα, τις τροπολογίες τους. Πράγματι είχαμε μια πάρα πολύ ενδελεχή συζήτηση και καταλήξαμε σε καλές ε, συμβιβαστικές προτάσεις που είμαι βέβαιος ότι βελτιώνουν το κείμενο δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Απλώς θέλω να τονίσω τα κέρια μηνύματα τα οποία θα πρέπει να παρουσιάσει αυτό το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμώσει τη θέση της στο πολυμέρα σύστημα. Και μάλιστα γρήγορα, μέσα στο διεθνές περιβάλλον. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παίξει το πρώτο ηγετικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, θα πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει μέσα σε ένα πολυμερές πλαίσιο σωστά και γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον, τη μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα ασφαλείας γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δυναμώσει το ρόλο της και, να συντονισ... το, το, συντονισμό της μέσα στο σύστημα Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας πιο αποτελεσματικής συμμετοχής στην, ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη Γενική Συνέλευση. but... Η Γενική του, του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη πολιτική τα χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τονίσουν το ρόλο τους στις πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα μέσα για να ενδυναμώσουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Τέλος, ε, χρειαζόμαστε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία θα ε, υιοθετήσει σαφή βήματα και δράσεις που θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό παίκτη στη διεθνή γεγονότα. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω και στους εκπροσώπους αλλά και στην Αντιπρόεδρο να παρουσιάσει μια τέτοια στρατηγική. Όσον αφορά τώρα τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, πιστεύω ότι είναι καλές. Είμαστε πρόθυμοι να τις υποστηρίξουμε Τώρα όμως στην τροπο, τροπολογία 7 όπως ζητούμε από τα κράτη-μέλη να μειώσει την εκπροσώπηση εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, θέλω να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία. Η τροπολογία 84 από, από τον κύριο William Monroe είναι σωστή. Η συγγήτρια λέει ότι η θέση της ε, ομάδας πιστεύει... Ε, βασίζεται στο πόσο αποτελεσματικές είναι. Εντάξει, δεν λέω, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ε, ρεαλιστι, πόσο ε, ρεαλιστικά λειτουργούν οι ομάδες. Την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούκαν. Ο κύριο Σάκε. Ως ε, ε, εκπρόσωπος του Σκιώδους Λάμστορ. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους άλλους συναδέλφους εξ ονόματος των φιλελευθέρων και την συμπερίληψη πολλών από των σκέψεών μας. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα και θα θέλαμε να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτη, Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορέσουν να βασιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και ιδιαίτερα σε καιρούς δημοσιονομικής ε, λιτότητας. Και τη στιγμή που ε, μπορούμε να δράσουμε ως παγκόσμιος παίκτη, υπέρ των πολιτών, αλλά και ο συνάδελφος Κούκαν το έθιξε αυτό. Δεν είμαστε υπέρ του εθνικισμού και του προστατευτισμού. Άρα αυτή η έκθεση, από αυτή την έκθεση μπορούμε να αντιλήσουμε διδάγματα. Να δούμε τι προκλήσεις έχουμε για το μέλλον και να αποτελέσει τροφή για σκέψη για το πώς θα πρέπει να ε, δράσουν και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δράσουμε ως παγκόσμιος παίκτη μέσω αποτελεσματικότητας και συντονισμού. Είναι μια δήλωση λοιπόν που σχετίζεται με την εν γέννη συνεργασία μας και ελπίζουμε να περάσουμε έμπρακτα σε πράξεις. Ευχαριστούμε κύριε Σάκε. Σόλτς, έχετε το λόγο. Σκιώδης από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε στα αγγλικά ο κύριος Σόλτς, αλλά και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για τη δουλειά της και για τη φροντίδα να συζητήσει με τους κοιόδησίτες. Εγώ διερωτώ με, γιατί μιλώ και εξ ονόματος της ε, Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ε, έγιναν πολλές τροπολογίες τις οποίες απορρίπτεται. Είστε υπέρ της τροπολογίας 11 μεν της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ίντα. Αλλά εγώ εκπλήσωμαι γιατί μιλάτε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς ε, οργανισμούς και συμμετοχή της ιδιότητα μέλους ε, στον ΠΟΕ της Ένωσης πέρα από τα κράτη-μέλη με αυτόν τον τρόπο έχουμε και κάποια ευθύνη να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα αμοιβαία κατανόησης, αλληλοαναγνώρισης των εμπορικών μας εταίρων. Έτσι, αμοιβαίας ε, ισοτιμίας, για να το πω έτσι. Και θα ζητούσα να μας εξηγήσετε γιατί προτείνετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόλτς. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις τελικά σχόλια παρακαλώ από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Α, υπάρχει κάποιο κάποιος άλλο. Με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Έχετε το λόγο. Μίλαν Μαν. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι θα πρέπει να σταθώ σε δύο δικές μου τροπολογίες που δεν αποτελούν αντικείμενο συμβιβασμού, αλλά θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα προς τις ε, διάφορες πολιτικές ομάδες και την εισηγήτρια. Η 135 για τον ε, ΟΑΣΕ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει θέση του παρατηρητή. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει δρόμο από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τον κανονισμό φαίνεται ότι ο Βαν Ρομπόι μπόρεσε να παρέμβει σε ε, διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς συναντήσεις Ευρωπαία. όπως την περίπτωση της Αστάνα πριν από την Βελγική Προεδρία και αυτό δεν είναι αρνητικό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το στάτους του παρατηρητή όμως δεν αναγνωρίζεται στον ΟΑΣΕ. Ως προς τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Θα πρέπει να μελετηθεί αυτό το θέμα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να οριστεί το στάτους του παρατηρητή σε όλους τους ε, ε, διεθνείς οργανισμούς και γι' αυτό έχω υποβάλει μια τροπολογία υπό αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Έχετε το λόγο, κυρία Μούνιθ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια. Ως προς την 135 και το περιεχόμενο δεν είναι ότι δεν θέλησα να τη λάβω υπόψη, αλλά πιστεύω ότι το θέμα του παρατηρητή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παρατηρητή, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουμε κατά μία βαθμίδα. Δηλαδή Πρέπει να δούμε πού μπορεί να γίνει πραγματικά μέλος και πού θα έχει το στάτους του παρατηρητή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε στον κανονισμό αυτό των οργανώσεων κατά πόσο μπορεί να έχει το στάτους του παρατηρητή ή όχι και θα το δω και στα πλαίσια του της τροπολογίας 135 ως προς το ΝΑΤΟ πιστεύω ότι θα πρέπει να ανέλθουμε κατά μία βαθμίδα ως προς την ε, συμμετοχή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κύριε Σόλτς, σε σχέση με τις τροπολογίες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, σκεφτούμε και να λάβουμε υπόψη ότι αναφερόμαστε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ, όπου όταν μιλάμε για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κανονισμό, δεν μπορούν να ενταχθούν αυτά τα θέματα στα πλαίσια αυτού του κανονισμού ή όταν μιλάμε για κράτη-μέλη που ορίζουν μια συγκεκριμένη στρατηγική. Πρόκειται για κρατικά αιτήματα και όχι και δεν αποτελούν, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ως προς την υπαριθμόν ένα, ένα, την, ένα μέρος της 4 και της 11 νομίζω ότι λαμβάνουμε υπόψη την άποψη της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου γιατί πρόκειται για συστάσεις για το πώς μπορεί να ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς και σε αυτή την περίπτωση στο ΠΟΕ και στις συναφείς οργανώσεις όπως η UNCTAD για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε τις πολιτικές που προωθούν αυτές οι οργανώσεις. Θα υπερψηφίσουμε, μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες που προανέφερα μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε μία συνολική άποψη και θα αναθεωρήσω τον κατάλογο ψηφοφοριών όπως σας είπα τώρα με τις αλλαγές που σας ανέφερα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Μούνιθ. Όπως γνωρίζετε θα ψηφίσουμε αύριο στην ΑΦΕΤ και τον Μάιο στην περίοδο συνόδου θα ψηφίσουμε την έκθεση. Το επόμενο θέμα προβλέπει μία συνάντηση και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό θα ήθελα οι υπάλληλοι που δεν έχουν άδεια να αποχωρήσουν, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες. Πριν προσέλθει η κυρία Γιάννα Ιμπάσκοβα, η οποία προβλέπεται να έρθει τώρα volete lasciare lasciare l'aula, ci prepariamo. Σας παρακαλώ να αποχωρήσετε τώρα για να προετοιμάσουμε την επόμενη συνάντηση και κλεισμένων των θυρών.